το μεσημέρι θα έχουμε την ψηφοφορία σχετικά με την έκθεσή του. Τώρα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχουμε την κοινή συζήτηση για τέσσερα, τέσσερις εκθέσεις, μακροοικονομική χρηματοδοτική ε, συνδρομή, πρώτα έκθεση Βίταλ Μορέρα, έκθεση ε, Μόρισλα Βαράνστοφ και η έκθεση Βίνκλερ. Καταρχήν θα έχουν το λόγο οι, οι και καταρχήν ο κύριος Μορέρα Μορέιρα για τέσσερα λεπτά. Κύριε Μορέα, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λόγο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας απευθύνω χαιρετισμό και να σας διαβιβάσω τον ενθουσιασμό μου στην ε, συμμετοχή αυτή, αυτού του σώματος που εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω σήμερα δύο εκθέσεις σε σχέση με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία και στην Αρμενία έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ισοζύγιο πληρωμών και το εξωτερικό χρέος αυτών των δύο χωρών του Καυκάσου. Μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, οι δύο αυτές χώρες επλήγησαν ε, στεναρά. Στην ε, περίπτωση της ε, Γεωργίας, η επίπτωση της κρίσης αφο, ε, επιδεινώθηκε μάλλον από τις άμεσες και έμεσες συνέπειες της ε, περσινής στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Ρωσία τον Αύγουστο του 2008 που ε, οδήγησε σε άμεσες και έμεσες ζημίες καθώς και σε εσωτερική μετακίνηση μέρους του πληθυσμού. Επίσης, επιδεινώθηκε η κατάσταση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και από το γεγονός ότι η Γεωργία και η Αρμενία εξαρτώνται από τον, τη μεγάλη γείτονα χώρα από το βορρά. Πρόκειται για μια δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση. Γι' αυτό οι δύο αυτές προτάσεις μακροοικονομικής έκτακτης χρηματοδοτικής συνδρομής θα μειώσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού και θα εξηγιάνουν το ισοζύγιο πληρωμών της Αρμενίας και της Γεωργίας. Γι' αυτό οι δύο αυτές εκθέσεις εγκρίνουν την ανάγκη επέκτασης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Αρμενία και τη Γεωργία. Και στα πλαίσια της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ζήτησα από τους συναδέλφους να εγκρίνουν αυτές τις δύο εκθέσεις χωρίς ε, τροπολογίες μέσα στα πλαίσια της απλοποιημένης διαδικασίας δύο αυτές εκθέσεις υποβάλλονται λοιπόν τώρα στο Κοινοβούλιο, αλλά θα θέλαμε να στυλιτεύσουμε την καθυστέρηση της Κομισιόν και του Συμβουλίου, ενώ γνώριζαν ότι θα έπρεπε τάχιστα να προωθήσουμε αυτή την μακροοικονομική χρηματοδοτική έκτακτη συνδρομή. Με αυτή μας λοιπόν τη θέση, δεν θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε επιφυλάξεις και ανησυχίες σε σχέση με τις συμφωνίες που προτείνονται. Και μερικοί από εμάς, εάν είχαμε άλλες εναλλακτικές λύσεις, θα υποβάλαμε τροπολογίες σε σχέση με ορισμένα κριτήρια που διέπουν την αρρωγή και συνδρομή αυτή για να βελτιώσουμε την διαφάνεια της διαδικασίας. Τώρα θα τελειώσω κυρία Πρόεδρε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα εγκρίναμε αυτές τις δύο συμφωνίες σε σχέση με τις δύο αυτές χώρες. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι άμεση στρατηγική σημασία σε αυτές οι δύο συμφωνίες μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και θα ήθελα να τις εγκρίνετε και τις δύο. μέσα στα πλαίσια της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής συνδρομής έκθεσης, εκθέσεις χωρίς τροπολογίες και οι δύο, το ξανατονίζω. Λοιπόν, επόμενος ο μιλητής είναι ο κύριος Ράνστοφ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε μια συζήτηση στην Επιτροπή για αυτή την έκθεση ε, προτείναμε μια απλουστευμένη διαδικασία εφόσον πρόκειται για θέμα που επήγει ιδιαίτερα. Αναφέρομαι στο η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή Δία στα Βαλκάνια και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα η οποία και εκείνη επιθυμεί να προσχωρήσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτή τη στιγμή υπάρχει αστάθεια οικονομική, υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, η χώρα ε, ε βρίσκεται ακόμα υπό την επίρρεια των γεγονότων του παρελθόντος υπάρχουν ακόμα πρέπει να, ε, ε, να επισκευαστούν οι καταστροφές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι θα σε Σερβία από άλλες περιοχές των Βαλκανίων και η τρέχουσα οικονομική κρίση οπωσδήποτε δεν συνέβαλε στη, δεν βοήθησε την κατάσταση. Οι βομβαρδισμοί μείωσαν την, τη γεωργική παραγωγή πέρσι την εποχή της συγκομιδής προέκυψαν ε, προβλήματα ιδιαίτερα σοβαρά για τη χώρα. Γι' αυτό κρίνω ότι είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τη βοήθεια στη χώρα αυτή και να ώστε να ξεκινήσει τις αρχές του επομένου χρόνου. Έχουμε λοιπόν για το λόγο αυτό προτείνει μια πλουστευμένη ε, ταχεία διαδικασία η οποία θα ωφελήσει τόσο τη Σερβία όσο και τις γειτονικές της χώρες που δεν ανήκουν στην, ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Κροατία που θα ήθελαν να γίνουν μέλη, αλλά και χώρες που ήδη ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πιθανώς να απειληθούν από αυτή την αστάθεια όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία ή η Βουλγαρία. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις χώρες αυτές και στην ευρύτερη περιοχή τους και για να βοηθήσουμε ειδικότερα τη Σερβία, προτείνουμε, όπως σας είπα, να εγκριθεί αυτή ε, η ταχεία απλουστευμένη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Σογκόρ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχω την τιμή να ε, σας παρουσιάσω την Επιτροπή Διεθνούς ε, την, ε, την, άποψη, την άποψη της, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η οικονομία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης έχει επηρεαστεί από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η Βοσνία Ερζεγοβίνα επέβαλε λοιπόν αίτηση για βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν πρότεινε να παρασχεθεί με τη μορφή δανείου 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα, ε, θα χορηγηθεί στο 2010 σε δύο δόσεις. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση ή όχι. Σύμφωνα με τις κανόνες της ισχύουσας συνθήκης, θα μπορούσαμε να πούμε γιατί να μην περιμένουμε να τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και να υποβάλουμε μια τροποποιημένη ε, διαδικασία και πρόταση. Ε, παρόλο την, το, το γεγονό ότι όταν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας το έργο μας θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Πιστεύω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να δείξουμε πολιτική δέσμευση και ε, ε, ευαισθησία και να δώσουμε τώρα τη βοήθεια στις χώρες των Βαλκανίων που τη χρειάζονται και όχι στις αρχές του επομένου έτους. Πρέπει και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε τόσο πολύ χρονικά την παροχή αυτής της βοήθειας πιστεύω. Γι' αυτό η Επιτροπή μας προτείνει η πρόταση παροχή βοήθεια στη Βοσνία Ερζεγοβίνη να εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Αβώνα, χωρί τροποποίηση, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία. Οι ε, συνάδελφοι τη Επιτροπή μα υποστήριξαν αυτή την πρόταση και ζητώ τώρα να την υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο επίτροπο κύριος Κάλλα. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σημειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την θετική και επικοδομητική στάση του Κοινοβουλίου σχετικά με την υιοθέτηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για τέσσερις χώρες, τη Γεωργία, την Αρμενία, τη Σερβία και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Έχουμε ε, υιοθετήσει ε, μία ε, μία μεθοδολογία που θα επιτρέψει εφόσον δεν υπάρχουν τροπολογίες να προχωρήσουμε ήδη από αύριο και ε, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες αυτές εντός των υπομένων και να εφαρμόσουμε τα προγράμματα που έχουμε καταρτήσει. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι ένα μέτρο επιλύσεως των κρίσεων και ε, χρηματικής συνδρομής είναι ένα μέτρο που έχει προβλεφθεί ε, για τις χώρες αυτές, για την Αρμενία, τη Γεωργία, την Βοσνία που έχουν πληγεί ε, την κρίση πάρα πολύ ε, λόγω των χρηματοοικονομικών τους δομών και της οικονομικής εξελίξεώς τους. Χρειάζεται λοιπόν προγράμματα τα οποία θα βοηθηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προσφέρει μακροοικονομική συνδρομή σε χώρες που καλύπτουν τα κριτήρια και όσον αφορά το μέλλον τώρα της συνδρομής αυτής σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας η οποία προβλέπει μια διαδικασία για μακροοικονομική συνδρομή με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής και του Συμβουλίου. Βεβαίως ε, θα χρειαστεί μακροπρόθεσμα να υπάρχει μια διεργασία συνεργασίας μεταξύ ε, των διαφόρων θεσμικών οργάνων που δεν ε, συνάδει με τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι είναι πολύ βασικό να εξετάσουμε πώς θα προχωρήσει στο μέλλον η χρηματοοικονομική συνδρομή στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις στο μέλλον θα μπορέσουν να διεκπεραιώνονται καταρχήν ταχαίως και αποτελεσματικά για να αντεπεξέλθουν της κρίσεως καλύπτοντας όμως τις ε, επιταγές της συνθήκης της Λισαβόνας ε, στα πλαίσια της διαδικασίας κοινής λήψης αποφάσεων διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά είναι χρήσιμα και εξετάζει τις τεχνικές πτυχές αυτών των θεμάτων στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας διότι μπορούν να προσφέρουν πολλά προτερήματα μέχρι όμως υιοθετηθούν αυτές οι διατάξεις το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποφασίζεται κατά περίπτωση περίπτωση είναι από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, όπως έγινε στην ε, πρόσφατη πρόταση Επιτροπής ε, για την Ουκρανία και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύντομα θα μπορέσουν να συμφωνήσουν και θέλω επίσης να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει μία αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών για την μακροοικονομική συνδρομή κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν αυτά τα θέματα γρήγορα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα ερχόμαστε τους ομιλητές εν ονόματι των πολιτικών ομάδων όπου πρώτα έχει το το λόγο ο κύριος Κουτάς εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την δουλειά τους και να πω και να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και τη Σερβία, συνδρομή που έρχεται σε πολύ σημαντική στιγμή για τις χώρες αυτές. Μετά από τα προβλήματα και τη δυστυχία της δεκαετίας του 90 και τις τόσες θεματοχυσίες έχει αρχίσει η διαδικασία της ανασυγκρότησης χώρες αυτές που σταμάτησε όμως λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης με ψηλά ποσοστά ανεργίας. Οι επενδυτές για το λόγο αυτό έχουν περιορίσει τις ε, παρεμβάσεις τους και τις επενδύσεις τους σε πολλές ε, χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Σερβία, η οποία επηρεάστηκε σοβαρά από την κατάσταση αυτή και γι' αυτό χρειάζεται, έχουν αυξηθεί ανάγκες της για εξωτερική μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. οι κοινωνικές και οικονομικές ε, ε, και προοπτικές της χώρας είναι πολύ δυσμένες, τα ποσοστά ανεργίας θα, δεν πρόκειται να μειωθούν σύντομα από ό,τι φαίνεται. Η οικονομική κρίση έπληξε τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι προτάσεις για μακροοικονομική χρηματοδυτική συνδρομή είναι ευπρόσδεκτες και αναγκαίες προκειμένου να σταθεροποιηθεί μια περιοχή η οποία πέρασε από πολλές δυσκολίες και παραμένει ακόμα ιδιαίτερα ευάλωτη. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των χωρών που θέλουν να ενταχθούν το συντομότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να λάβουμε ε, επίσης υπόψη. Γι' αυτό επήγει η παροχή βοήθειας προς τις χώρες αυτές. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν ε, την, ε, και να, τη χρηματοδοτική συνδρομή το ταχύτερο δυνατό χωρίς να ε, ξεκινήσουμε συζητήσεις για διαδικαστικά θέματα και να περιμένουμε την έγκριση και την έναρξη εφαρμογής της συνθήκης Λισαβόνας. Ο επόμενος ομιλητής δεν παρίσταται, άρα το λόγο έχει ο κύριος Κόβαλ για το ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Αμάδα των Συντηρητικών. Ευχαριστώ. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ευθύνονται για την κατάσταση στη Γεωργία και γι' αυτό καλό θα ήταν στο, ψήφισμα αυτό να αναφέρουμε ότι η κατάσταση πριν ε, από το 2008 ήταν πολύ καλή και η διαμάχη το 2008 οδήγησε σε αυτή την ε, επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ε, και στο μέλλον καλό θα ήταν η χώρα αυτή να έχει τη δικιά της προοπτική προς την Ευρώπη. Θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση στο Κάφκασο, η οι διάφορες κυρώσεις δεν επιτρέπουν η γεωργία να αναπτυχθεί φυσιολογικά και γι' αυτό και πρέπει να τονίσουμε ότι η γεωργία θα έπρεπε να επωφεληθεί αυτή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για να μπορέσει να αναπτυχθεί οικονομικά ε, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της και αυτή η ενίσχυση θα έπρεπε ίσως να ενισχυθεί, να αυξηθεί. Άρα το ερώτημα εδώ είναι να φροντίσουμε η συνδρομή αυτή να φτάσει στη Γεωργία ήδη εντός του 2009 και η, ε, οι ε, διαδικασικές λεπτομέρειες δεν πρέπει να εμποδίσουν να φτάσει η βοήθεια αυτή το 2009 εις ε, την ε, Γεωργία και ε, θα έπρεπε επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι το πρόγραμμα του Καυκάσου δεν έχει υλοποιηθεί και ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η σχέση μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσίας θα διεκπαιρεώνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τώρα ερχόμαστε στους ε, επόμενους ομιλητές ε, και πρώτος είναι ο κύριος Πορέβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καθίσταται σαφές ότι η προτινόμενη μακροοικονομική συνδρομή για την ε, Γεωργία, Αρμενία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σερβία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν αρκούν όμως και εδώ λαμβάνω υπόψη ιδιαίτερα την κατάσταση της ε, Γεωργίας η οποία θα λάβει αυτή την οικονομική αρρωγή που δεν θα επιλύσει πολλά προβλήματα. Μιλάμε για 65 και 35 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε όμως τι συνέβη ως προς την ε, ε, σύραξη με τη Ρωσία. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Ε, θεωρώ ότι τα 100 εκατομμύρια δεν επαρκούν. Γι' αυτό για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας θα πρέπει να αποφασιστεί και η διαφοροποίηση προμήθειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν δεν τους δώσουμε την δυνατότητα ανάπτυξης, θα το κάνει αυτό η Ρωσία. Και ξέρετε ποια είναι τα συμφέροντα που διέπουν αυτή την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή. Καλή πρόταση της Επιτροπής, αλλά ως προς την χρηματοοικονομική συνδρομή δεν αρκεί. Ευχαριστώ. Για τη διαδικασία Catch the Eye δεν βλέπω να υπάρχει καμία αίτηση λόγου, άρα τον λόγο έχει πάλι ο κύριος Επίτροπος Κάλλας. Έχετε τον λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονίας η οποία σε μεγάλο βαθμό μπορεί να παράσχει κοινωνική υποστήριξη και συνδρομή σε χώρες της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ομόφωνα υποστήριξαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει τις γειτονικές χώρες. Κάποιο αξιότιμος βουλευτής είπε ότι αυτή η διαδικασία τα διαδικαστικά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν το έργο μας, αλλά υπάρχουν οι διαδικασίες όμως που πρέπει να τηρηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην τήρηση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόζονται και να τηρούνται σαφείς κανόνες κατά την παροχή συνδρομής, χρηματοδοτικής συνδρομής και στο εγγύς μέλλον θα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συμφωνία πλαίσιο η οποία θα καθιερώσει ένα ειδικό πλαίσιο για την παροχή τέτοιας χρηματοδοτικής συνδρομής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη στιγμή, βεβαίως θα αποφασίζουμε, αυτή μέχρι τώρα ε, αποφασίζουμε ε, χωριστά για κάθε περίπτωση με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις που είναι μια από τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν, αν υπάρξει ένας μηχανισμός ε, ταχείας λήψης αποφάσεων, οπωσδήποτε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα μας επιτρέπει και αυτός ο μηχανισμός θα μας επιτρέψει να παρέχουμε τη βοήθεια στις χώρες που τη χρειάζονται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα έχει και, έχουν και πάλι το λόγο να δευτερολογήσουν οι συγητές και καταρχήν ο κύριος Μορέιρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εκφράσω τρεις ε, τελικές ε, σκέψεις. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή χρειάζεται διότι έχει πολιτική σημασία. Είναι θέμα γοήτρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθά αυτές τις χώρες στα πλαίσια της σχέσης καλής γειτονίας. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά πολιτικά και κοινωνικά αυτές τις χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να δράσουν δημοκρατικά και να παγιώσουν το δημοκρατικό τους πολίτευμα. Η αρρωγή αυτή, η χρηματοοικονομική αρρωγή θα πρέπει να τηρεί δύο όρους. Να ανταποκρίνεται στις ε, εξαιρετικές ε, χρηματοοικονομικές δυσκολίες και οι χώρες αυτές να μην χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για άλλους λόγους, δηλαδή για στρατιωτικές ε, δαπάνες ή σκοπούς. Θα ήθελα να υποστηρίξω το γενικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση χρηματοοικονομικής αρρωγής και γι' αυτό θεωρώ ευπρόσδεκτο το συμβασμό του Επιτρόπου Κάλλας ε, για αυτό το θέμα και ελπίζω η επόμενη Επιτροπή να σταθεί στο ύψος αυτού του ε, συμβιβασμού και να φτάσουμε σε ένα γενικό κανονισμό που να διέπει την χρηματοοικονομική αρρωγή. Ευχαριστώ. Τώρα πάλι ο κύριος Ράνσοφ για δύο λεφτά και αυτός. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ένας μεγάλος συγγραφέας είπε κάποτε ότι τα Βαλκάνια είχαν, ανελάμβανε περισσότερες ιστορικές ευθύνες από αυτές που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για τον Κάφκασο, διότι και οι λαοί της περιοχής αυτής ανέλαβαν περισσότερες ιστορικές ευθύνες από αυτές που μπορούσαν να χειριστούν και να αντιμετωπίσουν. Και ίσως ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε τις χώρες αυτές, να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Διότι χωρίς τα Βαλκάνια δεν είναι ολοκληρωμένη η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Σέρβοι αστευόμενοι είπαν ότι μόνοι φίλοι τους είναι οι Έλληνες και ο Θεός, πρέπει να τους δείξουμε ότι υπάρχουμε και εμείς και υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και, το... και τώρα ο κύριος Σόμπορ πάλι για δύο λεφτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, και οι τέσσερις χώρες για τις οποίες σήμερα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή την χρειάζονται λόγω της κρίσεως γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βγουν από την κρίση και για τη γεωργία η βοήθεια των 46 εκατομμυρίων η οποία θα ενισχύσει την αποκατάσταση της χώρας αυτής μετά από την κατάρρευση των οικονομικών οικονομικών της ε, ε, με την ε, κρίση με τη Ρωσία. Βλέπω ότι για την Αρμενία αναφέρονται 100 εκατομμύρια για την ε, ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης, την επίλυση των προβλημάτων και την χρηματοδότηση του ελλείμματος. Η Σερβία η οποία έχει πληγεί σοβαρά επανέρχεται ε, εις την τάξη και είναι μια ενδεχόμενη υποψήφια χώρα σε συμφωνία συμφωνία σταθερότητας και γι' αυτό πρέπει να βοηθηθεί πολιτικά. Η Βοσνία τεγοβινη είναι επίσης μια δυνητική υποψήφια χώρα ε, για συμφωνία συνδέσεως και γι' αυτό προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να την συνδράμει. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνω πρέπει να εκδηλώσουμε την πολιτική μας δέσμευση να δώσουμε στις χώρες αυτές τη βοήθεια που χρειάζονται τώρα αντί να μακρηγορούμε συζητώντας την ε, χωρίς λόγο. Για την ομάδα του ΕΛΚ εγώ προτείνω η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για τις χώρες αυτές θα πρέπει να υιοθετηθεί τώρα και ζητώ από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την πρότασή μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ε, ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Αξιότιμοι συνάδελφες, σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε ε, σύντομα την συνεδρίαση διότι θα αναλάβει ε, την Προεδρία ο Πρόεδρος